Voilà, je vous propose de, de commencer. Et donc on commence par euh, un vote. Donc on... Ας αρχίσουμε και αρχίζουμε μια ψηφοφορία. Μια και μόνη λέει ο Πρόεδρος. Οπότε να σας αφήσω ακόμα ε, λίγη, λίγη ώρα για να καθίσετε. Λοιπόν, αρχίζουμε την ψηφοφορία για την ε, έκθεση, την γνωμοδότηση της κυρίας Ορφσκοκ, ενίσχυση οικονομικής, κοινωνικής και δαφικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θα ήθελα να καθίσει ο κύριος Λένας. Meneer Ολλανδικά. Έχει eh? eh? έρθει η ώρα τη ψηφοφορία, κύριε Λέναρτ, λέει στα Ολλανδικά ο πρόεδρο. Πάμε. Ψηφίζουμε λοιπόν. Συμβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Υπέρ. Κατά άποχες εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε την τροπολογία 51 σε τρία τμήματα. Τμήμα πρώτο, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το θέλετε έλεγχο παρακαλώ, ας το επαληθεύσουμε. Είναι το πρώτο τμήμα της παραγράφου 51. Περισσεύει ένας από το ΕΛΚ. Της τροπολογίας 51, όχι παράγραφο. Συγγνώμη. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα καταπίπτει. Το τρίτο τμήμα υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται και το τρίτο. Η τροπολογία 63 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα καταπίπτει και συμβιβαστική 6 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Η τροπολογία 38 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται που είμαστε τώρα 45 υπέρ κατά απόχες. Νομίζω ότι χρειάζεται παλήθευση αυτό. Παρακαλώ, ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 48 είπε Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 49 επε. κατά αποχές απορρίψετε 50 επε. κατά αποχές εγκρίνεται 52 επε. κατά αποχές εγκρίνεται 53 επε. κατά αποχές εγκρίνεται 54 επέ. κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 64 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 68 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 75 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 76 σε τρία τμήματα, τμήμα πρώτο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά απόχες για να το ελέγξουμε αυτό παρακαλώ πέρασε 23-21 εγκρίθηκε ε, το τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 79 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ή, ορίστε. Έλεγχο θέλετε για την 82. Παρακαλώ, επαληθεύουμε την 82. Άρχιτε η ψηφοφορία. Πέρας. Ισοψηφία. Τι έγινε. Ναι. Pour Δυστυχώς, για την ηλεκτρονική ψηφοφορία δεν γίνεται. Δεν είναι ηλεκτρονική ψηφοφορία αυτό, επαλήθευση είναι. Δεν είναι ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πρόεδρε, δεν θεωρείται ηλεκτρονική ψηφοφορία. Επαλήθευση είναι ηλεκτρονική. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι δεν ψήφισε βουλευτής που ήταν ε, παρόν ή παρούσα, διότι δεν έχει την κάρτα. I'm συγγνώμη, αλλά ψηφίσαμε. Δεν ήταν σαφές. Ζητήσαμε επαλήθευση και η αξιότιμη βουλευτής θα έπρεπε να σταματήσει την ψηφοφορία και να πει ότι δεν έχω την κάρτα μου και τα λοιπά. Τελείωσε, τώρα πάει. Το τσεκάραμε, προχωρούμε. Ζητώ συγγνώμη, αλλά ως πρόεδρος επιμένω ότι έχει απορριφθεί. Η τροπολογία 83, ψηφί υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 1. Τι, μέσα 83 θέλετε έλεγχο. Πάμε. Non, c'est la même chose. Πάλι το ίδιο θα γίνει. Πέρασε. Απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Μητροπολογία 6 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Η συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. Η τροπολογία 16 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. Η συμβαστική 4. Τσεκ για τη 16 λοιπόν, ελέγχουμε τη 16. Άρχεται η ψηφοφορία και τελειώνει. Απορρίπτεται. Συμβαστική 4 Ειπέ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 είπε, Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 27 είπε, Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση που αρχίζει τώρα. Le vote Εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια.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 Θα Σας άφησα λίγες στιγμές έτσι για να μπορέσετε να φύγετε όσοι θέλετε να αποχωρήσετε. Okay, Καλώς. Θα σας πρότεινα να περάσουμε στο σημείο 9 της μερισσές διάταξής μας. Σας παρακαλώ. On peut commencer? Merci. Μπορούμε να αρχίσουμε. Ωραία. Στο σημείο 9 τη ε, ημέρης της διάταξης έλεγα έχουμε την παρουσίαση μελέτης με θέμα την ένταξη των προσφύγων στην Ελλάδα, την Ουγγαρία και την Ιταλία. Θα δώσω μέσω στο λόγο στην κυρία Μανουέλε Σαμέκ για ένα τέταρτο για να μας παρουσιάζει τη μελέτη της. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αυτή η μελέτη παρουσιάζει μια συνολική έποψη για την ε, εξέλιξη της ε, πολιτικής μας όσον αφορά την ε, υποδοχή και ένταξη σε Ιταλία, Ελλάδα και Ουγγαρία των προσφύγων. Να δούμε τι είναι τελευταία τριετία, να δούμε πώς οι ζωές είχαμε και τι πολιτικές φυρμόστησαν σε αυτές τις τρεις χώρες και που αναεφίσανται σημαντικά προβλήματα, να δούμε τι έγινε με την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και επίσης να δούμε το πώς όλα αυτά επηρέασαν την κοινή γνώμη. Και το μεταστευτικό και το προσφυγικό επομένως. Οπότε ε, έχουμε εδώ πέρα ανάλυση διαφόρων εκθέσεων αναχώρα και, και ένα κείμενο αναλυτικό, desk analysis. Ποιος μιλάει εκτός μικροφώνου. So I came here as a Hungarian MEP to... Εγώ είμαι εδώ, είμαι Ουγγαρέζα Ευρωβουλευτής και ήρθα εδώ για να ακούσω τα, τις σχετικές εκθέσεις με ενδιαφέρει, αλλά παρακαλώ κύριε Πρόεδρε, μπορείτε να επιβάλλετε την τάξη, γιατί εδώ πέρα ο κόσμος συμπεριφέρεται σαν σε καφενείο. Κάνουν πάρα πολύ θόρυβο και γίνεται, γίνεται χαμός, οπότε είναι αδύνατο κανείς να ακούσει τι λέει η ομιλήτρια. Παρακαλώ Πρόεδρε, επομένως, ζητήστε από τους συναδέλφους να περάσουν έξω, να θέλουν να πάνε στην ε, καφετερία και εκεί να τα πούνε και να αφήσουν τους ενδιαφερόμενους να ακούσουν. Manifestement, ils le font. <laughs> Madame, à uh, So... Έχετε το λόγο κυρία. Και τώρα, ε, μια που δώσετε μόνο 15 λεπτά, θα σας παρουσιάσω εν συντομία τα βασικά συμπεράσματα αυτή τη συγκριτική έκθεση και στη συνέχεια επίσης να δούμε τις αναχώρα εκθέσεις ε, όπως αυτά υπάρχουν στο website. Πρώτον, αυτές οι ισροές για αυτές τις τρεις χώρες. Υπάρχουν κάποιες νομιότητες μεταξύ αυτών των χωρών ε, όσον αφορά τη θέση τους στις διαδρομές των μεταναστών, αλλά ε, υπάρχει τελείως διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά την ένταξη και όσον αφορά την υποδοχή και των ασύλων και των μεταναστών και, και των πρόσφυγων. Οπότε από το 2014-2015 έχουμε πάρα πολύ μεγάλες αυξήσεις οι οποίες θα είναι αναπάντεχες και επίσης σε αυτές τις χώρες δεν υπήρχε προηγουμένη σοβαρή εμπειρία όσον αφορά την ε, υποδοχή και την ένταξη των των ασύλων και των πρόσφυγων. Οπότε ε, αυτές οι τρεις χώρες είναι χώρες τράνζιτ, ε, διέλευσης και όχι χωρίς προορισμού, γιατί ο κόσμος έφτασε σε αυτές τις χώρες και κατόπιν προσπαθούσε να μεταβεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, περιοχής Ευρώπης, βορειότερα. Οπότε ό, με όλα αυτά διαπιστώνει ότι έχουμε ε, αυξανόμενο ρυθμό και ποσοστό απόρριψης. Οπότε πέφτει ο μέσος όρος όσον μεσο όρο οσον αφορα την πρωτοβάθμια λήψη απόφαση για τις αιτήσει ασύλου. Τώρα να ρίξουμε μια σύντομη ματιά το πώς έχει κατάσταση κάθε μία από αυτέ τι χώρες. Ε, αυτά που σας ε, ανέφερα προηγουμένω είναι κάποιε ομοιότητε. Υπάρχουν και κάποιε διαφορές. Η Ελλάδα είναι το βασικό σημείο εισόδου όσον αφορά την Ανατολική Μεσοσογειακή Διαδρομή. Το 16 και το 17 ήταν ε, μεταξύ των πρώτων ε, χωρών της Ένωσης όσον αφορά τις αιτήσει ε, ασύλου σε σχέση με τον πληθυσμό και ήταν πάνω από το διπλάσιο του μεσόρου των 28. Τώρα η σύνθεση των ετούντων ε, διαφέρει σε σχέση με τις άλλες δύο χώρες που εξετάζουμε γιατί είχαμε πολύ περισσότερες γυναίκες και ανηλίκους είτε νεότερους των 18. Μιλούμε για το σχεδόν 40% σε σχέση με το 32% που ήταν ε, ο μέσος όρος Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό διότι οι πάρα πολλοί από αυτούς που έφτασαν ε, και ζήτησαν άσυλο προέρχονται από την ε, Συρία και κυρίως από έχουμε ε, το 16 πάρα πολλές οικογένειες. Επίσης έχουν πάρα πολλούς ασυνοδεύτους ανηλίκους οι οποίοι είναι μικρότερο ποσοστό των, των, ανηλίκων, των ανηλίκων σε σχέση με το μέσο όρο των 28 για το 16 η, το ποσοστό αναγνώρισης το 16 το 2016 ήταν κάτω από το 24% σχέση με το σχεδόν 61% της Ένωσης που είναι ο μέσος της όρος. Ουγγαρία. Ήταν, ήταν το βασικό σημείο η εισόδου όσον αφορά την διαδρομή των Δυτικών Βαλκανίων και ε, η κορυφή, το μάξιμου των ε, τήσεων έφτασε το 2015 που ήταν η χώρα αυτή με τη μεγαλύτερη εισρωή από τους 28 ε, όσον αφορά τις ε, αιτήσει και ήταν ε, περίπου 40% του συνόλου των αιτήσεων στην Ένωση των 28 και είχαμε πάρα πολλά περιστατικά είχαμε όσον αφορά τώρα Τη αιτήσεις είχαμε 18 αιτήσει για κάθε χιλίου κατοίκου και στη συνέχεια όταν έκλεισαν τα σύνορα σε αυτή τη χώρα ε, έπεσε ο αριθμός των αιτουμένων άσυλο από 177.000 πήγανε στις 29.000 μετά και ε, τώρα στις 4.000 σχεδόν. Επομένως, πολύ μεγάλη μεταβολή. Σε αυτή την περίπτωση μεγαλύτερη ομάδα των ε, ε, Ισραηλόντων, των, αυτών που φτάνουν εκεί από το Αφγανιστάν και τη Συρία. Άρα μεγάλη διαφορά σε σχέση με τη σύνδεση αυτών που πάνε στην Ελλάδα. Το 2016 στην Ουγγαρία έχουμε το χαμηλότερο ποσοστό αναγνώρισης, 8,4% μόλις. Γιατί όπως θα θυμάστε είχαμε 60,8% για την Ευρώπη των 28. Ιταλία, και πάλι έχουμε εδώ μεγάλε διαφορέ από τι άλλε δύο χώρε. Το βασικό σημείο εισόδου αφορά τη διάδρομο, τη διαδρομή τη κεντρική Μεσογείου. Και το, το, το υψηλότερο σημείο ήταν το 16 και το 17 για τις αφήξει. Και πρόκειται για την δεύτερη χώρα μετά από την Γερμανία όσον αφορά τον αριθμό των ετούντων πέραν του ποσοστού επί του πληθυσμού βέβαια, γιατί η Ιταλία έχει μεγαλύτερο πληθυσμό από τις υπόλοιπες δύο χώρες που μελετούμε και στην Ιταλία επίσης έχουμε ε, πάρα πολλούς ε, ασυνοδεύτους ε, ανήλικους για την Ευρώπη των 28. Οι περισσότεροι που φτάνουν εκεί προέρχονται κυρίως από την Αφρική, ιδίω από την Ιγυρία Και πολύ περισσότεροι είναι από ό,τι στις άλλες δύο χώρες σε σχέση με το σύνολο της Ευρώπης των 28. Είναι ενήλικες νέοι μεταξύ 18 και 34 ετών και το 85% εξ αυτών είναι άντρες. Και θυμηθείτε ότι στην Ελλάδα έχουμε 40% γυναίκες. Άρα τελείως διαφορετική είναι προκειμένου η σύνθεση. Τώρα ο μέσος όρος του ποσοστού αναγνώρισης του 16 ήταν υψηλότερος από στις άλλες δύο χώρες. 39% ε, Πάλι όμως υπολείπεται πολύ από τον Ευρωπαϊκό Μεσόρο. Πώς τώρα προχώρησαν και εξελίχθηκαν οι πολιτικές όσον αφορά την ένταξη και την υποδοχή. Θυμηθείτε σε αυτές τις τρεις χώρες έχουμε τις χώρες, ε, τις βασικές χώρες ε, ε, άφηξες, επομένως κυρίως είχαμε μέτρα, μέτρα υποδοχής και όχι τόσο ένταξης. Οπότε είχαμε βέβαια ποικιλία προσέγγιση για αυτές τις τρεις χώρες. Κυρίως η Ιταλία, αλλά σε μικρότερο βαθμό η Ελλάδα προσπάθησαν να βελτιώσουν τα συστήματα υποδοχής και ένταξης, ούτω ώστε να αναβαθμίσουν τις σχετικές τους υπηρεσίες, εγκαταστάσεις, να απλουστεύσουν τη διαδικασία της ε, αναγνώρισης και όλα τα σχετικά με τις αιτήσει, οπότε οι αιτούντες άσυλο να αναγνωριστούν, τότε να μπορούν να ψάξουν δουλειά και να ενταχθούν όσο γίνεται ταχύτερα ε, Επίση, ιδίως στην Ιταλία. Άλλαξε η προσέγγιση και προσπαθήσαν να εμπλακούν περισσότερο οι περιφερειακές και δημοτικές αρχές, περισσότερο από ό,τι πριν. Τώρα εμπλέκονται επομένω οι τοπικές αρχές στην υποδοχή και ένταξη. Τελείως διαφορετική προσέγγιση της Ουγγαρίας μετά από τη μεγάλη αύξηση του 2015 που θυμάστε ήταν πρωταθλήτρια η χώρα της ε, Ισραήλ κλείσαν τα σύνορα, βάλανε τον φράχτη και κόψανε την ε, δημόσια επιδότηση στήριξη κόπηκε η δημοσιοκρατική χρηματοδότηση. Οπότε τα περισσότερα από τα μέτρα υποδοχή γίνονται από τι ΜΚΟ. Αν τώρα ρίξουμε μία ματιά ει του στα τα στοιχεία που αφορούν την ε, διεθνή σύγκριση για τι πολιτικέ τις μεταναστευτικέ, είναι τα πράγματα εδώ αντιπροσωπευτικά. Μπορεί να δείτε ότι το 2014 η Ιταλία ε, ήταν λίγο παραπάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης των 28 και η Ουγγαρία και η Ελλάδα κάτω από το μέσο όρο. Όμως, αφήνουν τώρα κάποια προβλήματα όσον αφορά τα μέτρα της ένταξης, κυρίως τότε περιορισμένες εμπειρίες που είχαν αυτές οι χώρες, ιδίω η Ελλάδα, αλλά και η Ιταλία. Όσον αφορά τη διαχείριση των ευξημένων εισρωών, των των και των προσφύγων. Οπότε και προσέξαν σε προβλήματα όσον αφορά την καθυστέρηση της καταγραφής. Ήταν πάρα πολλοί αυτοί που ερχόντουσαν. Οπότε υπήρχε δυσκολία στη διαχείριση όσον αφορά την καταγραφή επίσης. Και η Ιταλία και η Ελλάδα δεν είχαν ε, τόσο στεγανή διοικητική δυνατότητα. Ούτε υπήρχε συνεργασία των εμπλεκομένων υπηρεσιών για την υποδοχή των, των άσυλων και των προσφύγων. Ε, the lack, the shortage. άλλο πρόβλημα ήταν ότι δεν υπήρχε χώρος, δεν υπήρχαν εγκαταστάσεις φιλοξενίας των των ε, άσυλων των προσφύγων και επίσης δεν είχαν γίνει σοβαρές επενδύσεις όσον αφορά την ένταξη στην αγορά εργασίας. Ε, και αυτό βέβαια διότι η Ελλάδα και η Ιταλία ήταν οι χώρες που κυρίως χτυπήθηκαν από την χρηματοοικονομική κρίση. Οπότε εκεί η αγορά της απασχόλησης πάσχει. Υπάρχει πρόβλημα για όλο τον κόσμο εκεί πέρα. Οπότε εκεί η ένταξη γίνεται ακόμη πιο δύσκολη. Έλλειψη επομένω χρημάτων. Άλλο πρόβλημα. Οπότε είχαμε όλο ένα και πιο αρνητική στάση του κόσμου προς πρόσφυγες και του άσυλο. Επίσης, εξετάστηκε μια που θέλαμε να δούμε τι διαθέσιμη ύλη υπήρχε, τα υλικά, τέλος πάντων το κόστος της πολιτικής ένταξης, Οπότε καταλήξαμε στο ότι σε αυτές τις χώρες βραχυπρόθεσμα ήταν ε, πολύ υψηλό το δημοσιονομικό κόστος για την υποδοχή. Πάντως, μακροπρόθεσμα όσον αφορά την ένταξη, το κόστος μάλλον είναι χαμηλότερο από ό,τι στις χώρες προορισμού. Εκεί που γίνονται κυρίως οι πολιτικές ένταξεις. Επίσης, το δου νου του έχει κάνει κάποιες μελέτες και κατέκτησε ότι υπάρχει απότομη αύξηση όσον αφορά το βραχυπρόθεσμο κόστος σε σχέση με το ΑΕΠ σε σχέση πάντα με τον προπαγωγό μέσο όρο τώρα. Χρηματοδότηση, το βασικό ταμείο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για αυτές τις χώρες είναι το Ταμείο ΑΜΙΦ το οποίο χρησιμοποιείται στην πρώτη φάση της διαδικασίας ένταξης στη ΔΕΗ, Ιταλία, φορά, στη, στη του συστήματος ε, υποδοχής και στην Ουγγαρία για παιδεία, ε, μαθήματα γλώσσας, ε, κατάρτισης, μέτρα κοινωνικής ένταξης για τους ανεγνωρισμένους. Στην Ελλάδα πάντως προσέκρουσαν σε προβλήματα υλοποίησης εκτέλεσης αυτών των ε, απορρόφηση αυτών των κονδυλίων. Πάντα σε επίπεδο υποδοχή και ένταξη. Επίσης, επιστρατεύθηκε το Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό Ταμείο, το Ταμείο Επενδύσεων, και ιδίω στην Ελλάδα, ούτω ώστε να υποστηριχθούν οι πιο μακρόπινε προοπτικέ ένταξη, ιδίω όσον αφορά την παιδεία, την επαγγελματική κατάρτιση, την απασχόληση, πολιτικέ κατά των διακρίσεων. Όμω, όσον αφορά το Κοινωνικό Ταμείο, το πρόβλημα είναι ότι δεν στοχεύει συγκεκριμένα του ζωντανού άσυλου και του πρόσφυγε, αλλά προβλέπει μέτρα για τους μειονεκτούντες. Οπότε έτσι καλύπτονται και οι τούντες και οι πρόσφυγες. Όπως σας προείπα, υπάρχουν προτείνοντας χώρε χώρες εκείνες από πλευράς της ε, συμπεριφοράς του κόσμου όσον αφορά τους ετούντες και τους ε, ε, πρόσφυγες. Το πρόβλημα της σε κάποιες χώρες υπάρχει συγκέντρωση αυτών των προσώπων σε κάποιες ε, περιοχές κοντά στα σύνορα, στην Ιταλία ας πούμε, σε κάποιες περιοχές της Νοτιού Ιταλίας, στην Ελλάδα. Επίσης ε, κυρίως έχουν συγκεντρωθεί αυτοί οι άνθρωποι στα νησιά. Στην Ουγγαρία είναι τα σύνορα με τη Σερβία. Οπότε το ότι έχουμε τόσες πολλές αφήξεις σε κάποια περιορισμένη συγκεκριμένη περιοχή αυτό παροξύνει την κατάσταση όσον αφορά την αρνητική στάση του κόσμου. Και βέβαια υπάρχουν κάποιες πολιτικές δυνάμεις ε, ευρωπαϊκές και εχθρικές στους μετανάστες που την κατάσταση την χειροτερεύουν. Οπότε, ε, είπαμε ότι έχουμε και κάποια στοιχεία από το Ευρωβαρόμετρο έρευνα τέλος του 16 και οπότε είπαμε ότι ε, τα αρνητικά αισθήματα είναι ψηλότερα από ό,τι στο μέσο όρο, 80% στην Ουγγαρία, 70% στην Ελλάδα και 69 στην Ιταλία και στην Ιταλία μάλλον το, πράγμα πάει προς τα πάνω. Ε, οπότε αυτή η επιδείνωση όσον αφορά τη στάση του κόσμου και την άποψη σε επίπεδο πολιτικής έχει συνέπειες για αυτές τις χώρες, για τη συνοχή, αλλά επίσης θα πρέπει από το βαρόμετρο να συμπεράνουμε το ότι έχουμε όλο ένα και περισσότερη άποψη, αίσθηση του κόσμου ότι έχουν εγκαταλειφθεί στις τύχες τους όσον αφορά τη διαχείριση του προβλήματος. Επίσης, έχουμε αυξανόμενα ποσοστά τα οποία ζητούν για πιο δυναμική ευρωπαϊκή πολιτική για το μεταναστευτικό και ανάληψη ευθυνών από περισσότερο κόσμο. Τώρα οι άλλε προκλήσει, αλλά προβλήματα θα πρέπει να υπάρχει μικρότερη πίεση όσον αφορά τι παραμεθόρε περιοχέ και να υπάρχει περισσότερη κατανομή των ε, ετούντων αλλά και των ε, προσφύγων. Οπότε χρειάζεται να βοηθήσουμε αυτέ τι χώρε σε σχέση με το να έχουν περισσότερε δυνατότητε για αποτελεσματικά μέτρα και για αντιμετώπιση των ε, ανισοτήτων. Και επίσης υπάρχει και το πρόβλημα του πώς θα φρενάρουμε αυτή την ε, αντιμεταναστευτική στάση του κόσμου και πώς ο ιδιωτικός τομέας και οι κοινότητες θα εμπλακούν στην υποδοχή, στην ένταξη. Αυτά όσον αφορά τη συγκριτική ανάλυση χρειάζεται περισσότερη συντονισμό και συνεργασία μεταξύ των ε, θεσμικών οργάνων, των κρατών μελών, Ούτως ώστε να κάνουμε σωστή κατανομή των ετούντων και των ε, μεταναστών. Χρειάζεται διακυβέρνηση πολυεπίπεδη, τοπικές αρχές, περιφερειακές αρχές να βοηθήσουν, σημαντικό. Το θέλουν οι, οι τοπικές περιφερειακές αρχές. Και να βοηθηθούν να αποκτήσουν δυνατότητες σχετικά με αυτά. Επίσης, το κόστος ένταξης και το πώς θα γίνει πράξη συνειδητοποίηση του προβλήματος και να αντιμετωπίσω και το πρόβλημα τη συλλογής δεδομένων και της εποπτείας του τι γίνεται ε, σε κάθε επίπεδο εθνικό και τοπικό. Εδώ θα βάλω τελεία και ευχαριστώ να απαντήσω τις ρωτήσεις σας ή δυνατόν. Ευχαριστώ κύριε Σάμεκ. Ο κ. Κάζνα δεν είναι εδώ από πλευρά ΣΕΛΚ. Κ. Κόζα. Köszönöm Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστώ πολύ για τη μελέτη αυτή. Και καταρχάς να πω ότι προέρχομαι από μια χώρα η οποία ε, πλήττεται και είναι και αντικείμενο της μελέτης, η Ουγγαρία. Υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε παρερμηνίες γιατί συμπεριλαμβάνουν αρνητικούς χαρακτηρισμούς και δεν βοηθάνε όλα αυτά στη σημερινή μας συζήτηση. Γιατί το θέμα είναι κρίσιμο και σημαντικό και πιστεύω ότι θα πρέπει να το κρατήσουμε σε ένα νυφάλιο επίπεδο, να ξεκαθαρίσουμε ε, τους όρους. Ποιος είναι μετανάστης, ποιος είναι πρόσφυγας, ποιος είναι οικονομικός μετανάστης, ποιος είναι λάθρο μετανάστης. Ε, όλοι αυτοί οι ορισμοί ανακατεύονται μεταξύ τους, αναμειγνύονται. Για την Ουγγαρία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν έχω σταματήσει να το τονίζω και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνουμε διάκριση κάθε φορά. Ποιος είναι τι και να διευκρινίζουμε τους όρους και τις έννοιες που χρησιμοποιούμε. Ε, πρέπει να βοηθάμε τον κόσμο. Αυτόν όμως τον κόσμο που έχει δικαίωμα να ζητήσει άσυλο και προστασία βάσει διεθνών συμφωνιών συχνά. Η ουγγρική ε, μεταναστευτική πολιτική βασίζεται στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ουγγαρίας. Ξέρετε ότι η χώρα μας είναι σχετικά μικρή χώρα. Ε, και ακούσαμε τώρα για το κόστος της εσωμάτωσης και πόσο δαπανάει ο καθένας. Η Ουγγαρία μπορεί να δαπανάει λιγότερα από τα άλλα κράτη-μέλη για την ενσωμάτωση και την ένταξη των μεταναστών. Αλλά χρηματοδότησε μόνη τη το φράχτη στα σύνορα, ο οποίο φράχτης εξασφάλισε Ε, την ε, ομαλή διέλευση των μεταναστών. 800 εκατομμύρια ευρώ κόστησε ο φράχτης αυτός και δεν έδειξε αλληλεγγύη η Ευρωπαϊκή Ένωση και βοηθήσαμε και προστατεύσαμε ε, και τα άλλα κρατημέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το φράχτη αυτό να παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα η μεταναστευτική πίεση και ροή. Θέλω να τονίσω και πάλι ότι Είμαστε υπέρ της κανονικής τακτοποιημένης μετανάστευσης αξιοπρεπούς που απορρέει από διεθνείς συνθήκες και υπάρχει ένα πλαίσιο νομικό και νόμιμο. Όταν έρχεται ο άλλος νόμιμα στη χώρα και ζητάει άσυλο βεβαίως. Αυτή τη μετανάστευση εμείς την υποστηρίζουμε. Γι' αυτό θέλω να σας κάνω την εξής ερώτηση. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε. Η Ελλάδα γεωγραφικά είναι πιο κοντά στη Μέση Ανατολή αλλά δεν κάνουν αίτηση ασύλου στην Ελλάδα. Ε, λιγότερες αιτήσει κάνουν από ό,τι στην Κεντρική Ευρώπη και στην Ουγγαρία. Γιατί δεν κάνουν τις αιτήσει ασύλου στην ε, Ελλάδα και έρχονταν να κάνουν στην Ουγγαρία. Και πώς βρέθηκαν στην Ουγγαρία, πέταξαν. Δηλαδή η πρώτη έτσι ασύλου θεωρείται πρώτη χώρα εισόδου η Ουγγαρία, μα αφού ήταν η Ελλάδα η πρώτη χώρα εισόδου στην οποία έφτασαν οι πρόσφυγες. Και είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθείτε αυτή η διαδικασία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για μένα προσωπικά και για την Ουγγαρία και νομίζω ότι μιλάω ξενόματος όλων των συναδέλφων μου. Ήθελα να τα πω αυτά. Βεβαίω και θα πρέπει να προστατεύουμε τους ανθρώπους, αλλά εκείνου που έχουν δικαίωμα στην προστασία αυτή. Να διευκρινίσουμε τους ορισμού και τις έννοιες που χρησιμοποιούμε. Και ένα τελευταίο, με το οποίο δεν έχει ασχοληθεί καθόλου η μελέτη, καν. Είμαι πεπισμένο ότι τα προβλήματα θα πρέπει να τα λύνουμε στη ρίζα τους. Κάθε φορά εκεί που δημιουργούνται να λύνονται. Άρα να αντιμετωπίσουμε τα αίτια της μετανάστευσης. Μιλήσατε και για τις χώρες Βίσεγκρατ. Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία. Έχουν ταπανίσει πάρα πολλά χρήματα και επενδύσεις στις χώρες προέλευσης καταγωγής των μεταναστών για να βελτιώνεται η παιδεία, η οικονομία, για να παραμένουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες στις χώρες τους. Και ένα τελευταίο. Η συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε καμία περίπτωση δεν έχει ολοκληρωθεί. Αλλά είναι σημαντικό η ευελιξία να... Ε, μάλλον η να είναι ευέλικτη, δεν υπάρχει μία λύση. Δεν μπορεί κανείς να μετεγκαθιστά τους πρόσφυγες και τους μετανάστες σε ένα κράτος μέλος. Και μια τελευταία παρατήρηση. Δεν θα πω ότι συγκλονίστηκα ή ότι σοκαρίστηκα ή ότι έμεινα άναυδος. Αλλά βλέπουμε πάρα πολλούς νεαρούς ανθρώπους και παιδιά, ασυνόδευτους ανηλίκους και γνωρίζουμε από αξιόπιστες πηγές ότι αυτοί που, θεωρούν, που δηλώνουν ανηλικοί δεν είναι καθόλου ανηλικοί, απλώς ε, πλαστογραφούν τα στοιχεία τους για να λάβουν ένα συγκεκριμένο καθεστώς. Συνοψίζοντας λοιπόν πρέπει να επαναλάβω ότι χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε. μετανάστευση να είναι τακτοποιημένη, να είναι συντεταγμένη με προστασία των εξωτερικών συνόρων για τα προβλήματα να λύνονται εκεί που δημιουργούνται. Και ο κόσμος να μένει στα σπίτια του. Και αυτοί που πραγματικά χρειάζονται προστασία, πραγματικά να αναβάνουν τα πάντα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Κανείς για τους σοσιαλιστές. Ο κ. Καβέσομπον δεν είναι εδώ. Ρομπέρ. Ο κ. Μπονιφέρ. Μετά Ρομπέρ. Ο Ρομπέρ πρώτα. Ευχαριστώ που για την παρουσίαση της μελέτης. Άκουσα ενδιαφέρουσα. Ερώτηση έχω. Και έχω και κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτη ερώτηση. Έχουμε αριθμητικά στοιχεία για το κόστος των μέτρων υποδοχής προσφύγων και ποια είναι η κατανομή του κόστους, τι αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι αναλαμβάνουν τα κράτη. Από ό,τι κατάλαβα στην Ιταλία ήταν 85% ε, που πληρώνει η Ιταλία και 15% που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις τρεις χώρες που παραθέσατε όπου μιλάτε για αυτό το πρόβλημα, αναφέρεστε στο κόστος, έχετε όμως στοιχεία. Αυτό είναι σημαντικότατο. Για να δούμε ποιο είναι το μερίδιο της ευθύνης μας ή ανευθυνότητάς μας στο θέμα αυτό. Πιστεύω και θα αναφερθώ σε αυτό εν συνεχεία για τα θέματα της ενσωμάτωσης. Όσον αφορά όμως την υποδοχή αυτή καθεαυτή των προσφύγων, συμφωνούμε στο γεγονός ότι η υποδοχή, η άφηξη, η χώρα υποδοχής είναι ευρωπαϊκή ευθύνη, ακόμα και αν υπάρχουν χώρες που είναι περισσότερο χώρες υποδοχής από άλλες. Παραθέσατε παραδείγματα όσον αφορά τις χώρες που είναι κυρίως χώρες υποδοχής. Δεύτερον, σωστά λέτε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα κοινή γνώμη. Εγώ δεν ανήκω σε εκείνους που πιστεύουν ότι η κοινή γνώμη σφάλει. Ούτε ανήκω σε εκείνους που πιστεύουν ότι έχει απόλυτα δίκιο κοινή γνώμη. Εν πάση περιπτώσει, Αυτά τα θέματα είναι θέματα ασύγνωστα, τα γνωρίζουμε ως αιρετοί εκπρόσωποι που μας θέτουν σε αντιπαράθεση την κοινή γνώμη. Συμφωνώ με αυτό που είπε ο Ούγκρος συνάδελφος. Ένα από τα προβλήματα, δυσκολίες που έχουμε σε αυτή την κοινή γνώμη είναι το εξή. Μιλάμε για άφηξη των προσφύγων. Δεν ξέρουμε. Μιλάμε άφηση προσφύγων για την αποδοχή, τη χορήγηση καθεστώτος ασύλου ε, των προσφύγων όταν εξετάζεται η κατάστασή τους για την ενσωμάτωσή τους ή αν μιλάμε πιο γενικά για θέματα μεταναστευτικά. Και πιστεύω ότι η κοινή γνώμη βλέπει ότι επικρατεί και μεγάλη σύγχυση. Για την κοινή γνώμη επικρατεί η ιδέα ότι υπάρχει ένα φαινόμενο παγκόσμιο μετανάστευσης, γενικό, που δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Και συγχαίουμε κάπως τα πράγματα. Και σε σχέση με το θέμα των προσφύγων όπου τίθεται ένα θέμα συστήματο αξιών. Αξιών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, θεμελιωδών δικαιωμάτων προ σεβασμό. Το θέμα τη μεταναστεύσεως είναι εντελώ διαφορετικό που παραπέμπει σε θέματα ισορροπίας μεταξύ των πληθυσμών που ίσω αφιχθούν και δυνατότητα ενσωμάτωση. Χρειάζονται εργατικά χέρια, διαφορετικέ ανάγκες σε κάθε κράτος εργατικών χεριών. Σχετικά με αυτό, στη μελέτη σας διάβαξα το γαλλικό κείμενο της σύνοψης, η τελευταία φράση που παρουσιάζεται λέει να ενθαρρύνουμε το συλλογικό πνεύμα και να ευαισθητοποίηση ε, όσον αφορά τα ωφέλη της μεταναστεύσεως. Δεν συζητούμε αυτό σήμερα. Το θέμα δεν είναι αυτό να εξετάσουμε τα ωφέλη της μετανάστευσης. Αλλά όταν μιλάμε για τους ε, πρόσφυγες που το θέμα των προσφύγων είναι εντελώς διαφορετικό. Ξέρουμε ότι είναι δυσχερέστατο ζήτημα διεξάγονται συζητήσεις εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η χρηματοδότηση της υποδοχής προσφύγων και της ενσωμάτωσης αυτών, έστω και προσωρινής, δεν ξέρω την της τάξη μεγέθους και της χρηματοδοτήσεως ε, εγκαταστάσεως ε, ε, σήματοχμευμάτων και φρακτών. Δεν μπορεί να είναι παρόμοια η αλληλεγγύη ευρωπαϊκή για αυτούς τους δύο στόχους τύχη και ενσωμάτωση. Αυτό πιστεύω αυτοί που εξετάζουν το θέμα είναι ότι το θέμα πρέπει ανάντι να εξεταστεί. Όσον αφορά το θέμα των προσφύγων ή μεταναστεύσεως, η εκ ε, αντιμετώπιση δεν είναι ίδια. Όσον αφορά τη μετανάστευση εν γέννη, χρειάζεται ε, αναπτυξιακή βοήθεια. Όσον αφορά την υποδοχή των προσφύγων, έχουμε ένα άλλο πρόβλημα προς την αντιμετώπιση. Αυτό παραπέμπει στην αποδιάρθρωση των χωρών προέλευσης και ξέρουμε ότι εκεί οι ευθύνε είναι εξαιρετικά περίπλοκες. Κλείνοντας. Η δεύτερη ερώτηση. Η πρώτη ερώτηση ήταν όσον αφορά το κατανομή του κόστους. Η δεύτερη ερώτηση τώρα. Στις τρεις χώρες που αναφέρατε, που υποδέχονται πρόσφυγες, δεν τίθεται μόνο το θέμα της ενσωμάτωσης των αφιχθέντων και της ενσωμάτωσης των προσφύγων που αποκτούν δικαίωμα μόνιμο εγκατάστασης. Υπάρχει κάποια ανάλυση όσον αφορά μακροπρόθεσμα θέματα όποτε γίνεται, επιστροφής, κάποτε επιστροφής αυτών, να επανέλθουν στις πατρίδες τους. Για το θέμα των προσφύγων σε σχέση με χώρες σε εξαιρετική κρίση, δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα θέμα οριστικό και τελικό. Στον βαθμό που κάποιες περιστάσεις για κάποια ποσοστά των πληθυσμών ε, είναι διαφορετικά. Καταστρέφεται η χώρα προέλευσης, η περιοχή από την οποία προέρχονται. Και κάποια στιγμή όμως θα μπορούν να επιστρέψουν οι πληθυσμοί όταν αποκατασταθεί κάπως η κατάσταση. Όταν λήξει η κρίση η κρίση που απειλεί τη ζωή τους όταν τελικά θα έχει λήξει. Πώς μπορούν να πιστέψουν αυτοί. Ευχαριστώ κύριος Μπονιφάη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και το Τμήμα Πολιτικής για τη σημερινή παρουσίαση. Δυστυχώς είχα μια ομιλία σε άλλη επιτροπή και δεν άκουσα την παρουσίαση. Έλαβα όμως το κείμενο. Και σας ευχαριστώ για τη δουλειά σας. Έχω κάποια σχόλια. Αναμφισβήτητα, η ενσωμάτωση των προσφύγων στις κοινωνίες μας παραμένει κρίσιμο ζήτημα για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Είμαστε το μέσο σοβαρής καταστάσεως. Απαιτείται συνεχής προσπάθεια πολιτικής ύψης στο επίπεδο, κυρίως να ολοκληρωθεί το πακέτο, η μεταρρύθμιση του πακέτου ασύλου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και μπαίνουμε στις λεπτομέρειες όσον αφορά το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αν δεν δώσουμε στην πολιτική ένταξη των προσφύγων την κατάλληλη προσοχή, θα είναι το λάθο. Ήμουν εισηγητή σε αυτή την επιτροπή για την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση στην αγορά εργασία των προσφύγων και χαίρομαι που πολλά σημεία που ανέφερα εγώ στην έκθεσή μου τονίζονται και στη μελέτη σα, ξεκινώντα από την κυριαρχία της υπο... τα μέτρων υποδοχής από αυτά ενσωμάτωση λόγω ελλείψεω μακροπρόθεσμη στατικικής και υπαρκών πόρων και λόγω της κατεπίγουσας ανάγκης των προβλημάτων που αντιμετώπισαν οι τρεις χώρες. Δεν μας εκπλήσει το γεγονός που διαβάζουμε τις μεγάλες διαφορές της πολιτικές που εφάρμοσε η Ουγγαρία από τη μια πλευρά και η Ελλάδα και η Ιταλία από την άλλη. Αυτό αντικατοπτρίζει την ανάγκη ενισχύσεως των προσπαθειών για την εξέβρεση εύρυθμου ευρωπαϊκού συστήματος που δεν θα μπορεί να εφαρμόζεται κατά το δοκούν από κάθε κράτος μέλος. Κυρίως λόγω του διακυβεύματος που είναι η ζωή και τα δικαιώματα εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Και είναι σαφές ότι αυτό αποτελεί θέμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και όχι μεμονωμένου κράτους μέλους. Επίσης, Φαίνεται προφανέ ότι τα συστήματα υποδοχή και ενσωμάτωση αυτών των χωρών εξαρτώνται απόλυτα από τη χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω κυρίως το ΑΜΙΦ και το ESF. Το τελευταίο δεν έχει σαν στόχο κυρίως τους ετούντες άσυλο. Το Κοινοβούλιο ζήτησε να διατεθούν κατάλληλοι επιτόπιοι πόροι αποτελεσματικά και γρήγορα. Χρειαζόμαστε το ESF να τονωθεί. Χρειαζόμαστε το ταμίφ Πρέπει να βελτιωθούν οι συνέργειες μεταξύ των άλλων πόρων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και να μην έχουμε σποραδικές και τυχε πρωτοβουλίες. Θέλουμε συνεκτική πολιτική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως αυτή τη διαδικασία. Πρέπει ε, να έχει τη συμμετοχή τοπικής περιφερειακή αυτοδιοίκηση και ενδιαφερομένων κύκλων κοινωνία των πολιτών που πολύ συχνά εφαρμόζουν τα προγράμματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το επεξεργόταν αυτό και προσβλέπουμε στο νέα πρόταση πολιτού δημοσιονομικού πλαίσιου για ισορροπημένη προσέγγιση όσον αφορά τα σχετικά θέματα. Επίσης, να προσθέσω κάτι, ότι πάντα υπάρχει ένα θέμα πολιτικής ευαισθησίας. Είναι δυσχερέστατο οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές και οι πολιτικά εκλεγμένοι εξωματούχοι να λάβουν δύσκολες αποφάσεις περί κατανομής πόρων του ΙΕΣΕΦ για προγράμματα που αφορούν την ενσωμάτωση των προσφύγων αντί για άλλες ευάλωτες ομάδες. Άρα πρέπει να υπάρχει ισχυρός σχεδιασμός και όθηση από πλευράς Ευρωπαϊκής ιδεμή, η, τα βραχυπρόθεσμα εκλογικά κίνητρα για την κάλυψη ευαλώτων ομάδων που ψηφίζουν, ε, διακύβευμα εκεί είναι πολύ ψηλό. Πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα, να δούμε που έγκυται το πρόβλημα. Ευχαριστώ για την έξοχη προσπάθειά σας θα είναι πολύ χρήσιμη για το έργο της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου. Επαναλαμβάνω, διότι σύντομα θα λάβουμε σημαντικές αποφάσεις περί σχεδιασμού διαθέσεως πόρων που είναι το κλειδί, το βασικό θέμα όταν συζητούμε τέτοια θέματα και αυτή είναι η άποψή μου και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κανείς για την ΚΟΕ, ούτε για τους πράσινους, ούτε το EFTD. Ο κ. Ντομίνικ Μαχτέν έχει λοιπόν το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία μου για την παρουσίαση της μελέτης που αφορά την ε, ένταξη, ενσωμάτωση των προσφύγων εις Ελλάδα, Ουγγαρία και Ιταλία. Χρησιμοποίησα τα αρχέτυπα χωρών για το φαινόμενο. Ευχαριστώ. Διότι ήσασταν ειλικρινείς όσον αφορά την ε, προσέγγιση της έκθεσής σας εύλογα τα στοιχεία. Υπάρχουν ελάχιστοι πρόσφυγες, κυρίως οικονομικοί μετανάστες υπάρχουν από ό,τι βλέπουμε. Ευχαριστώ. Αποδεικνύεται και το λέτε σωστά ότι είναι πύλες εισόδου. Συνεπώς χώρες διέλευσης. Εφόσον είναι λοιπόν χώρες διελεύσεως, δεν έχουν επιλογή. Είτε επιταχύνουν τις διαδικασίες καταγραφής νομιμοποίησης αυτών, ούτως ώστε οι μετανάστες να μπορούν να πάνε σε άλλη χώρα, άλλων προορισμών και θεώρησε ότι αυτό αφορά κυρίως την Ελλάδα και την Ιταλία, χρειάζονται πάνω σε αυτό προσπάθειες, είτε κλείνουν, κλειδώνουν. Και από ό,τι κατάλαβα αυτό ισχύει για την Ουγγαρία. Κάπου αλλού έχετε κάποια μεροληψία πολιτική θα έλεγα. Να επενθυμίσω ότι εδώ και δύο χρόνια για μια κρόαση είχαμε υποδεχθεί τον Ευρωπαϊκό πρόσωπο του Ερυθρού Σταυρού και πρόεδρο ενώσεως διεθνούς μεταναστεύσεως. Ο κύριος ήταν από την Αφρική, δεν ξέρω αν θυμάται πρόεδρος. Και ο κύριος αυτός μας εξήγησε ότι η μετανάστευση ετησίως αφορά 60 εκατομμύρια άτομα. Και εκείνοι έκαναν έρευνες. Και μπόρεσαν να αποδείξουν ότι από τα 60 εκατομμύρια, το 10%, 6 εκατομμύρια δηλαδή, είχαν σαν στόχο τις χώρες, τις ευρωπαϊκές. Ταυτόχρονος, ο Ερυθρός Σταυρός χρησιμοποιούσε την ίδια ρητορική όπως και εσείς και οι προλαλήσαντες. Αναφερθήκατε στην ένταξη, στην ενσωμάτωση. Ο Ιθός Σταυρός είχε τρεις προτεραιότητες. Η πρώτη, ενσωμάτωση. Η δεύτερη, εξέβρεση εργασίας. Και η τρίτη, πιο εκπληκτικό αυτό, οργάνωση της οικογενειακής επανένωσης. Αρκετά σημαντικό αυτό. Και απαντώ στον κύριο Ροσφόρ. Αν κάποια στιγμή Βλέπουμε το ενδεχόμενο να επιστρέψουν στις πατρίδες τους, οι πραγματικοί πρόσφυγες, που αντιπροσωπεύουν λίγους. Θα καταλάβετε ότι ο όρος ενσωμάτωση με ενοχλεί. Θα προτιμούσα τον όρο ε, απορρόφησης, αφομοίωσης, διότι θέλουμε να τους ενσωματώσουμε πάση θυσία με τα ε, έθιμά τους. Αλλά αυτό τους οδηγεί σε μια απομόνωση κοινοτική, κοινοτικοποίηση. Η κοινοτικοποίηση εκνευρίζει τους ντόπιου που έχουν παραδόσεις. Είναι παλιό αυτό. Αν πας στη Ρώμη πρέπει να, κάνεις, να ζεις όπως οι Ρωμαίοι. Δεν πρόκειται περί ενσωματώσεως, αλλά αφομοιώσεως. Και εκεί μεροληπτήσατε. Αναφερθήκατε σε κακές αντιδράσεις των πληθυσμών. Γιατί είναι κακή αυτή η αντίδραση. Είναι μια αντίδραση. Γιατί κακή. Γιατί αντίδραση ε, να είναι κακή. Μας το είπε ο Ούγγρος βουλευτής. Κάνει ό,τι μπορεί η Ουγγαρία με τα διαθέσιμα μέσα. Εκεί που βρίσκεται. Στη θέση που είναι. Είναι μια αντίδραση θεμητή. Αναφερθήκατε σε αντιευρωπαϊκά κινήματα. Δεν υπάρχουν αντιευρωπαϊκά κινήματα παρά μόνο άνθρωποι που διαπιστώνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τεχνοκρατική, άκρος τεχνοκρατική δομή παίρνει λάθος αποφάσεις. Και υφίσταται η Ευρώπη, αγαπητή κυρία μου. εχει χιλιά 1000-1500 χρόνια ιστορία, έχει παραδόσεις. Δεν υπάρχουν αντιευρωπαϊκά κινήματα Και τελικά τι κάνει. Ε, υπάρχει Ελλάδα. Δεν είναι ότι εφεύραν την Ελλάδα τώρα. Υπάρχει Ελλάδα και αντιδρά ο πληθυσμό. Η τεχνοκρατική δομή που εκπροσωπείται η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η επιτροπή που δεν εκλέγονται από κανέναν, εκείνοι στέλνουν κείμενα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για επικύρωση. Το ξέρετε. Έναντι αυτού αντιδρούν. Άρα είναι θεμητή η αντίδραση, αγαπητή κυρία μου. Εφόσον εσείς μας εξηγήσατε την μελέτη, ειλικρινά λυπούμε που θέτω τόσο με αυτόν τον τρόπο την ερώτηση. Αντί να περάσω από Ελλάδα, Ιταλία και Ουγγαρία, αν αυτοί οι άνθρωποι περνούσαν από το διαμέρισμά σας, από το σπίτι σας, θα χαιρόσασταν ή θα είχατε μια αντίδραση. Πιστεύω ότι θα είχατε μια αντίδραση θεμητή. Διότι το ψυγείο σας, διότι η κρεβατοκάμαρά σας, τα παιδιά σας είναι εκεί και πρέπει να αντιδράσετε εσείς σαν μητέρα της οικογένειας. Λοιπόν, η καταλάπηση, η καταπολέμηση της αρνητικής νοοτροπίας και να ζητηθούν ευρωπαϊκοί ε, πόροι που πρέπει να αυξηθούν. Αυτή είναι πάντα η λύση. Αύξηση, αύξηση. Τελειώνω, τελειώνω, Πρόεδρε. Νομίζω ότι μίλησαν 5 λεπτά, 7 λεπτά. Η αύξηση των πόρων, λοιπόν. Ποιο πληρώνει. Πού βρίσκονται τα χρήματα, από την τσέπη πιανού βγαίνουν. Πρέπει πάντα να προτείνεται λύση. Και συμφωνώ με τον Ούγγρο βουλευτή πάνω σε αυτό. Και το είπε και ο Ροσφόρ. Η πρώτη λύση είναι να αντιστραφούν οι μεταναστευτικές ροές. Δεν έρχονται για τα όμορφα μάτια μας αυτοί εδώ, έρχονται τις συμφέροντά τους. Όπως πηγαίνουν διάφοροι παραμεθόροι εργαζόμενοι και πάνε από τη Γαλλία στην Ελβετία να εργαστούν, γιατί παίρνουν περισσότερα χρήματα. Είναι εθνική προτίμηση. Είμαι Γάλλος ε, ε, βουλευτής στο Ευρωκοινοβούλιο, προτιμώ να στηρίζω τους Γάλλους. Λοιπόν, θα πρέπει να παραμείνουν στις χώρες προέλευσης οι πληθυσμοί του μέσω πολιτικής συνεργασία για την ανάπτυξη. Και καλύτερα παρά να αυξήσουμε τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και των διαφόρων ταμείων για να του ενσωματώσουμε και όχι να του αφομοιώσουμε, θα πρέπει όλε αυτέ οι επενδύσει να πηγαίνουν για την ανάπτυξη σε ευφυεί επενδύσει σε συνεργασία με τι ε, χώρε προέλευση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ολοκληρώσαμε τι ομάδε. Τι θέλουν να μιλήσουν. Παρακαλώ να προσπαθήσετε να μιλήσετε δύο λεπτά, διότι θα ήθελα η κυρία Σάμεκ να είναι σε θέση να απαντήσει. Παρακαλώ, κάντε μια προσπάθεια και ο Τόμας Μάν. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ είμαι Γερμανός. Και κάθομαι δίπλα σε έναν Ούγγρο, τον φίλο μου τον Άνταμ Κόσα. Αγαπητέ Άνταμ. Αν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε θα έλεγα μακάρι, αλλά το 2015 εμείς υποδεχτήκαμε τους πρόσφυγες που ερχόντουσαν από την Ουγγαρία. Και θέλω να πω ότι οι Ουγγρικές αρχές παρακάλεσαν τις Γερμανικές να δραστηριοποιηθούν και πληρώσαμε πικρό τίμημα γιατί ακούσαμε ότι έρχονται πάρα πολλοί και δεν ελέγχονται και πάρτε τους όλους. Εμείς είμαστε ε, περήφανοι για τον όρο ε, η κουλτούρα της ε, ε, υποδοχής, ότι είναι όλοι ευπρόσδεκτοι. Τώρα δεν είναι πια ευπρόσδεκτοι, λέτε. Ε, συμφωνώ ότι πρέπει να κάνουμε τη διάκριση. Ε, τούντες άσυλο, μετανάστες, πρόσφυγες, οικονομική μετανάστευση κλπ. Βεβαίως, δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι, δεν λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Τότε στο Κοινοβούλιο, εγώ στην έκθεση Μπενιφέη, ήμουν στη συζήτηση για την ένταξη των ε, προσφύγων στην αγορά εργασία. Ήμουν και σκιώδη συγητής μάλιστα από το ΕΛΚ. Εργαστήκαμε πολύ καλά σε αγαστή συνεργασία. Και... Ακούσαμε τις επιφυλάξεις από την ε, ε, θεμητή και νόμιμη αντίδραση. Τι ανοησίες είναι αυτέ, Κοιτάξτε τους ανθρώπους. Πώς ζουν, σε ποιες συνθήκες. Υπάρχουν πολλοί εθελοντέ που βοηθούν για να γίνει η ένταξή τους και η ενσωμάτωση στην κοινωνία και τους στηρίζουν. Και είναι σωστό. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τη ριζοσπαστικοποίηση. Ναι, σωστή, δίκαιη κατανομή, αλλά παρακαλώ και αλληλεγγύη στην κατανομή αυτή και να φροντίσουμε πραγματικά να μην ε, υπάρξει τώρα μια ιδιαιτερότητα των χωρών Βίσεγκρατ απέναντι στα άλλα κράτη-μέλη της Ένωσης. Να μην αφήσουμε αυτό να γίνει, δεν επιτρέπεται. Θα πρέπει να οικοδομούμε από κοινού και τις ποσοστώσεις από κοινού να τις ε, επομιζόμαστε και να τις επιμεριζόμαστε όπως και το κόστος. Αλλιώς δεν γίνεται. Ε, πολύ καλή μελέτη και πολύ χρήσιμη. Ναι στην αλληλεγγύη, ναι στην κοινή προσπάθεια και να μην ακούμε αυτά που λένε κάποια κρουπούσκουλα επειδή φωνάζουν περισσότερο από τους άλλους. Θα πρέπει να μπορούμε να ε, λέμε όχι στη ροζοσπαστικοποίηση και να βασιζόμαστε στην ελεγγύη. και αυτή γίνεται μόνο από κοινού. Δεν θα πρέπει να χτίζουμε νέους φράχτες αλλά να φροντίσουμε με τις ιδιαιτερότητες, μάλλον για τα κοινά να συζητάμε και να εργαζόμαστε με ε, τις πλειοψηφίες, με τις μειοψηφίες και όχι να μπλοκάρουμε. Έχω πάρα πολλά να πω. Τι να πω μέσα σε δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρεπέρο, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα, σας ευχαριστούμε κυρία για την μελέτη και την παρουσία της. 20 αιώνες από τότε που είχαμε κόσμο να σύρεται ως μόνο μάχος και εγώ ξέρω ότι τι άλλο σκλάβο στη Ρώμη. Πάνε όλα αυτά. Τώρα φτάσαμε το 2017-18 και ο κόσμος άλλαξε. Οπότε το πρόβλημά μου με την μελέτη είναι το εξή. Δεν είναι τόσο πρόβλημα. Είναι ότι το, το τα είπανε συνάδελφοι. Μπενιφέ, Ροσφόρ. Πρώτα-πρώτα είδαμε τι είναι τα τελευταία χρόνια με αυτέ τι τρεις χώρες. Απροσδόκητο 100%. Α, ε, μοναδικό. Ποτέ δεν είχαν αντιμετωπίσει τέτοια εισβολή μεταναστών, προσφύγων των Περθών και ήταν απροετοίμαστες. Ναι, λέμε και ξαναλέμε για την ένταξη. Είχαμε και την έκθεση Μπενιφέ που ήταν για την Άλντε ο σκιώδης. Αλλά όταν μιλούμε για υποδοχή ανθρώπων και την μεταγενέστερη ένταξη, αυτό σημαίνει πρώτα-πρώτα γνώση. Μα χώρες που δεν είχαν αντιμετωπίσει τέτοια πάντα στο παρελθόν, πού να τη βρουν τη γνώση, να τους έρθει μάνα ως μάνα εξ και από μεριά χρήμα. Και το θέμα είναι ότι τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μάλλον τη στιγμή που ζήτησε ελληνική από τα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμφώνω θα έπρεπε να επιδείξουν ελληνική. Όμως το θέμα είναι ότι τότε η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ήταν έτοιμη να πάει και να βοηθήσει αυτές τις χώρες. Τις ΜΚΟ, τις κρατικές αρχές, να βοηθήσει στην υποδοχή και κατόπιν να εξηγήσει τι ένταξη θέλουμε στην παιδεία, στην δημόσια υγεία. Πόσα λεφτά ανήλωσε για όλα αυτά τόσα χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρία Σόιντροβα. Σας ευχαριστώ. Που... Που το λόγο. Νόμιζα δεν... Ε, πραγματικά είναι άνθρωποι, δεν είναι αριθμοί και οι εγγύοι η αλληλεγγύη. Γίνεται λόγος για ένα κύμα μετανάστευσης. Ε, ποιο είναι το πρώτο πρόβλημα, η πρώτη προτεραιότητα για τους πολιτικούς, η ασφάλεια. Και δεν μπορώ να τη διαχωρίσω την ασφάλεια από την αλληλεγγύη. Θέλω να ευχαριστήσω για τη μελέτη, παρόλα αυτά, την οποία θεωρώ βάση για τη συζήτηση, αλλά τώρα χρειαζόμαστε επίκαιρα στοιχεία ενημέρωση. Έχει μεταξελιχθεί η κατάσταση. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Δεν είμαστε στο 17 πια. Θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ενσωματώσουμε τον κόσμο αυτόν στην εκπαίδευση, στην εργασία. Χρειάζομαι ε, στοιχεία από την Ελλάδα μαθαίνουμε ότι δεν πηγαίνουν πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Παραμένουν οι καταβλισμοί, παραμένουν τα διάφορα κέντρα υποδοχής τα οποία διαμένουν οι άνθρωποι αυτοί και ε, αδρανούν. Δεν φεύγουν, δεν εργάζονται, ε, δεν επιστρέφουν ε, στα σπίτια τους, δεν εκπαιδεύονται, δεν κάνουν τίποτα. Θα πρέπει οπωσδήποτε να το δούμε και με καινούργια στοιχεία. Τα στοιχεία που μας δίνεται εδώ είναι του 2014. Τι γίνεται με τα ε, αριθμητικά στοιχεία και τα στατιστικά του 2018. Η κατάσταση είναι πολύ πιο περίπλοκη από αυτό που μας δείχνει η μελέτη. Ευχαριστώ. Η κυρία Μορβάη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα κι εγώ να ε, μιλήσω και φοβάμαι ότι ο κύριος Τόμας Μαν παρεξήγησε και παρανόησε τόσα συνέβησαν το 2015. Ο κύριος Τόμας Μαν ως Γερμανός λέει ότι έκανε τεράστια χάρη στην Ουγγαρία ε, δεχόμενος ως Γερμανία ε, αυτά τα εκατομμύρια, εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες ήτανε. Αλλά εσείς τους προσκαλέσατε στην Ευρώπη. Η κυρία Μέρκελ, η καγκελάριος και η γερμανική κουλτούρα του καλωσορίσματος που βγαίνατε και με ταμπέλες και με πανό και τους καλωσορίζατε. Δεν τους κάλεσαν οι Ούγγροι στην Ευρώπη αυτούς τους ανθρώπους. Οι Ούγγροι υπέφεραν από την κατάσταση αυτή όταν ε, ήταν ε, στον Ανατολικό Σταθμό και κατέκλυσαν ε, τα τρένα μας στο Σέγκετ και σε άλλες πόλεις με στη νύχτα ξυπνήσανε ε, τους αγρότες, τις αγρότησες σε απομακρυσμένα μέρη, στην Ήπεθρο, στην επαρχία. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Δεν θα ξαναπάρουμε, δεν μας κάνατε χάρη. Εσείς τους προσκαλέσατε, πάρτε τους επιτέλους. Εμείς δεν θέλουμε να τους έχουμε στην Ουγγαρία. Αυτά που λέτε εδώ είναι σαν να λέτε αυτά που λέει αντιπολίτευση στην Ουγγαρία που θέλει να έρθει στα πράγματα στις 8 Απριλίου. Εσείς όμως χαίρεστε ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ακούγοντας αυτά που λέει ο κύριος Τόμας Μαν. Να σταματήσουμε λέει το βέτο, να μην είναι εμπόδιο πια η Ουγγαρία ε, στον δρόμο αυτό που θέλετε να χαράξετε και να συνεχίσετε με αυτή την αξιοθρύνητη πολιτική της μετανάστευσης που έχουν ε, αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Μέρκελ και την έχουν επιβάλει στην Ουγγαρία. Ελπίζω πραγματικά να είναι αρκετά σόφρονες οι Ούγγροι και να μην το επιτρέψουν αυτό να υλοποιηθούν αυτές οι προσδοκίες και ο Θεός να σώσει και να ευλογεί την Ουγγαρία. Να δώσουμε πέντε λεπτά στην κυρία Σάμεκ να απαντήσει. Ε, I'm really interested in this debate. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση και θέλω να σας τονίσω ότι μελέτη κάναμε. Δεν κάναμε κανένα είδου μανιφέστο ιδεολογικό, οπότε εξετάσαμε κάποια στοιχεία. Δεδομένα ότι, ότι ήταν διαθέσιμο και ξεκαθαρίσαμε ευθύ εξ αρχή το θέμα τη ορολογία για να ξεκαθαρίσουμε περί τίνους συζητούμε. Το θέμα ήταν η ένταξη των προσφύγων και είπαμε συγκεκριμένα ότι εξετάζουμε Ουγγαρία, Ελλάδα και Ιταλία. Και ήταν πάρα πολύ σημαντικό να γίνει η διάκριση μεταξύ των των άσυλων και των προσφύγων. Διότι ανεγνωρισμένοι πρόσφυγες δικαιούνται να διαμείνουν στην χώρα αφίξιος και επίσης έχουν δικαίωμα πρόσβασης η πάσα υπηρεσία διαθέσιμη στην λογοχώρα, διότι αν έχουν την αναγνώριση τη ιδιότητας του πρόσφυγος, ότι δηλαδή έχουν διαφύγει από πόλεμο, δίωξη τη οικογένειά του κλπ. αιτούντε άσυλο είναι άλλη περίπτωση. Υποβάλλουν την αίτηση αναγνωρίσεω, φάνουν σε κάποια χώρα και κατόπιν ακολουθείται μία διαδικασία στη χώρα αφήξεως για να εξεταστεί κατά πόσον ε, θα τους απονεμηθεί αναγνώριση ή ου. Παίρνει κάποιο χρόνο αυτή η διαδικασία και κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου χρειάζονται κάποιο είδους ε, στέγαση, πλαισίωση, οπότε εάν αναγνωριστούν τελικά τότε θα πρέπει να αναζητούν ε, μέτρα για την ένταξή του, αγορά απασχόληση κλπ. κλπ. Εάν κρατά πολύ αυτή η διαδικασία ε, μάλλον αυτή η διαδικασία που ακολουθεί την αναγνώριση, ε, δύσκολα εντό εργασία όμω μπορούν να κάνουν κάποια άλλη δουλειά, εθελοντέ, δάσκαλοι ξένη γλώσσα, τη γλώσσα του, τέλο πάντων διάφορες τέτοιες ε, πολιτικές. Αυτό θέλω να σας ξεκαθαρίσω, ότι είναι συγκεκριμένη η χρήση αυτών των όρων. Και σήμερα από ε, τη μελέτη ξεκαθαρίζουμε τι θα πει πρόσφυγες, τι θα πει τον άσυλο, τι θα πει μετανάστες εν γέννη, γιατί πολλές φορές δεν έχουμε γενικώ ό,τι στοιχεία χρειάζονται. Έχουμε μόνο γενικά και όχι ανά ομάδα των προσώπων. Τώρα, όσον αφορά το κόστος, ε, για κάποια μελέτη, επί τη βάση κάποιων συνεντεύξεων, οπότε δεν μπορούμε ακριβώς να υπολογίσουμε το κόστος υποδοχής και ένταξης στις ε, τρεις ε, αυτές χώρες. Απλώς εξετάστηκε τι στήριξε έλαβε χώρα από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, ευρωπαϊκά ταμεία. Τώρα, όσον αφορά τις ε, πολιτικές επιστροφής δεν αφορά τους πρόσφυγες, οι πρόσφυγες δεν μπορούν να γυρίσουν διότι διατρέχουν κίνδυνο σε περίπτωση επιστροφής. Άρα θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε περί τίνος ομιλούμε. Όσον αφορά τώρα την αρνητική στάση του κόσμου, δεν είπα κακή στάση, είπα αρνητική. Αρνητική όσον αφορά την αντίδραση αυτών που άπνιζαν στο ερωτηματολόγιο στην έρευνα και είπα ότι αυτό εξηγείται. Και είπα διότι οι χώρες αυτές ε, είχαν να αντιμετωπίσουν ε, εκτεταμένη εισρωή από μετανάστες. Και αυτό εξηγεί πόθεν αυτή η αρνητική στάση. Δεν κάνω αξιολογική κρίση. Είπα ότι είναι πρόβλημα και κάτι πρέπει να γίνει σχετικά με αυτό. Τώρα επίση, όσον αφορά την επικαιροποίηση των πληροφοριών αυτή, η μελέτη έγινε πέρυσι. Οπότε υπήρχαν αναστοιχεία μέχρι νομίζω Ιούνιο του 2017. Τώρα έχουμε στοιχεία μέχρι και μου φαίνεται αρχές του 18 για τις ε, αφήξεις και προκύπτει ότι οι αφήξεις μειώνονται. Όμως ακόμη είναι πολλοί αυτοί που έχουν υποβάλει αίτηση και περιμένουν την απάντηση, την αναγνώριση ή μη. Και βρίσκονται ακόμα σε αυτές τις χώρες. Το πρόβλημα με αυτούς είναι ότι μέχρι ότου ληφθεί σχετική απόφαση είναι ε, εκρεμής η, υπόθεση τους. Είναι σε κάποιο νομικό κενό, δεν μπορούν να δουλέψουν, τίποτα δεν μπορούν να κάνουν. Άρα θα πρέπει να προβληματιστούμε. Κάποιο είδους πολιτική θα πρέπει να εξεύρουμε ούτω ώστε να μπορέσουμε να τους ε, εντάξουμε σε κάποιο πρόγραμμα και τελικά να συμβάλλουν, να βοηθήσουν τις κοινότητες εκεί όπου ευρίσκονται. Αυτά δεν το βάζουμε τελεία. Ο πρόεδρος, σας ευχαριστώ κυρία. Η επόμενη μας είναι 27 Τρίτου στις 2.30 ώρα στις Βρυξέλλες. Ευχαριστούμε και τους Δερμήνες. Γεια σας.